Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσουμε παρά τις επαναλαμβανόμενες δυσκολίες της Δευτέρας, του απογεύματος της Δευτέρας. Ξέρω ότι δεν έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή ρύθμιση, αλλά ας αρχίσουμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ανταλλαγή απόψε με την αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής στην ε, EU Now for Atalanta και μετά θα ασχοληθούμε με τις δύο αποστολές στα Παλαιστινιακά εδάφη θα έχουμε μαζί μας τον εργό της αποστολής Μπαμ Ράφα, συνταγματάρχη Αλέα Φαγκράς και τον εργό της αποστολής Γιουροπούκολ. Τώρα, μεταξύ των μελών της unav έχουμε τον κύριο, την κυρία Νικολάη που δεν είναι εδώ και τον κύριο Ζαλόφσκι, στον οποίο αμέσω θα δώσω το λόγο αν θέλει να μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης. Αυτό. Ευχαριστώ. Λάβατε μια λεπτομερή έκθεση αναφορικά με την επίσκεψή μας ε, στο Τζιπούτι. Γραπτή έκθεση. Ως εκ τούτου θα σχολιάσω απλά εν συντομία. Από 13 μέχρι 15 Νοεμβρίου ε, έλαβε χώρα η επίσκεψη και οι συναντήσεις μας είχαν ως αντικείμενο τις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιχείρηση Αταλάντα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις αποστολές τροφίμων και την καταπολέμηση της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας. Κάναμε λοιπόν ε, συναντήσεις με τους επικεφαλείς των αποστολών χώρα η οποία είναι υπεύθυνη για την αποστολή είναι η Γαλλία. Συνδεθήκαμε με τον αρμόδιο άπαρχο και τους ε, αξιωματικούς του, αλλά και με εκπροσώπους των στρατευμάτων της Γαλλίας που είναι σταθμευμένα στο Τζιμπουτί, αλλά και εκπροσώπους αμερικανικών στρατευμάτων Επίσης με εκπροσώπους της κυβέρνησης του Τζιμπουτή, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, με υπουργούς της κυβέρνησης, με τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την αποστολή αυτή, για την αποστολή κατά της πειρατείας από πλευρά των τοπικών αρχών. Η εντύπωση που μας δόθηκε λοιπόν ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή, στον Ινδικό ωκεανό και στον ε, κόλπο. 25 σκάφη συμμετέχουν στις ε, επιχειρήσεις και δεν αποτελούν τις μοναδικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Επίσης, ε, συμμετέχουν αμερικανικές δυνάμεις αλλά και στρατεύματα του ΝΑΤΟ. Η συνεργασία δε μεταξύ των στρατευμάτων των διαφόρων χωρών είναι πολύ καλή και μας είπαν ότι είναι εξαιρετική η ανταλλαγή πληροφοριών. Δημιουργήθηκε επίσης στο κόλπο του Άντεν ένας ε, ασφαλής, ένας διάδρομος αν θέλετε ασφαλείας προστατευμένος από τον οποίο μπορούν να περάσουν με ασφάλεια τα ε, πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ωστόσο, υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μας ανησυχούν. Κατά πρώτον, παρά το γεγονός ότι από σήμερα ο κόλπος του Άντεν είναι αρκετά ασφαλής, οι επιχειρήσεις των πειρατών απομακρύνονται από τις ακτές της Σομαλίας προς Ανατολάς. Και σήμερα η κατάσταση είναι η εξή. Βρουν ακόμα και πιο κοντά στις Ινδικές ακτές παρά στις Αφρικανικές ακτές. Άρα το πρόβλημα ουσιαστικά δεν έχει επιληθεί, έχει απλά μετατοπιστεί προς Ανατολάς. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις, απλά έχουμε μετατοπιστεί προς την Ανατολή. Κατά δεύτερον, φαίνεται ότι οι πειρατές και είναι καλύτερα εκμεταλλευμένοι πλέον, αλλά και έχουν στη διάθεσή τους πιο καλό εξοπλισμό. Άρα, όλο και πιο συχνά έχουμε ανταλλαγή Έχουμε ε, ένοπλε σειράξει. Ε. Άρα, οι επιχειρήσει μας ως τώρα ήταν επιτυχής. Αλλά επειδή είναι τεράστια η περιοχή, ουσιαστικά απλά υπάρχει μία μετατόπιση του προβλήματος. Μιλάμε για μια ναυτική περιοχή η οποία καλύπτει έκταση μεγαλύτερη από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα της ε, επίσκεψής μας, της αποστολής μας, για να αποτελέσουν τη βάση μιας ε, συζήτησης. Να σας πω λοιπόν ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία εξεγάγαμε. Καταρχάς, συνειδητοποιούμε και την αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα της πειρατείας δεν μπορεί να επιληθεί χωρίς να επιληθεί πρώτα το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει συνολικά η χώρα της Σομαλίας. χωρίς να οικοδομηθεί ένα εύρυθμα λειτουργών κράτος. Και άμεση συνάρτηση αυτού είναι η υποστήριξη προς μία ε, προσωρινή ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας, η οποία de facto θα ελέγχει την, την περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η υποστήριξη λοιπόν προς την κυβέρνηση δίνεται από πλευράς της ε, Ουγκάντα κυρίως. Και ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο πιο ε, μεγάλης οικονομικής βοήθειας. Γιατί από πλευρά της Ουγκάντα η βοήθεια είναι στρατιωτικής φύσεως. Ένα άλλο εκρεμές ζήτημα σε ό,τι αφορά του, την εκπαίδευση των ε, συνοριοφυλάκων στην Σομαλία. Για τη δημιουργία ενός στρατού, ο οποίος θα μπορούσε με αποτελεσματικό τρόπο να ελέγχει το νότιο τμήμα της χώρας Επίσης, πολλά θέματα συνδέονται με την ενίσχυση της ε, οικοδόμησης, αν θέλετε, κρατικών δομών, θεσμών. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. η εντολή από πλευρά Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις ε, κατά της πειρατείας προβλέπει επιχειρήσεις ε, στην ξηρά αλλά και στη θάλασσα και η εντολή για την, για την ε, επιχείρηση Αταλάντα αφορά αποκλειστικά ναυτικές επιχειρήσεις. Ενώ είναι σαφές ότι τα κέντρα των πειρατών είναι στην ξηρά. Και οι δραστηριότητες αστυνόμευσης για να κατασχεθούν για παράδειγμα οι εξοπλισμοί των ε, πειρατών θα ήταν πάρα πολύ σημαντική, σημαντικό επιτεύγμα. Για πολιτικούς όμως σκοπούς και για πολιτικούς λόγους δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όμως να το εξετάσουμε στον δεχόμενο, να εξετάσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα ενδεχόμενων επιχειρήσεων επί ξηράς, σε ό,τι αφορά τη σύλληψη των πειρατών. Οι ναυτικές δυνάμεις οι οποίες ε, συμμετέχουν στην ε, επιχείρηση Αταλάντα έχουν τις ε, σχετικές δυνατότητες. Άρα έχουμε και τις τεχνικές και τις στοχευτικές δυνατότητες να ξεκινήσουμε τέτοιες επιχειρήσεις επί ξηράς. Είναι όμως πολιτικός πώς ευαίσθητο το θέμα. Ωστόσο, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αξίζει τον κόπο να το κοιτάξουμε ως ενδεχόμενο. Κάτι άλλο. Η μεγαλύτερη ενίσχυση προς ένα κέντρο εκπαίδευσης στο Τζιμπουτί, όπου θα καταρτίζονται, θα εκπαιδεύονται οι συνοριοφύλακες. Η επιχείρηση Αταλάντα έχει να κάνει με την αρρωγή και τη συνεργασία με τις Σομαλικές Αρχές. σε ό,τι αφορά και την προστασία της ακτογραμμής. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθεσε και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Τσιμπούτι είναι το εξής. Στο Τσιμπουτί τα έσοδα προέρχονται από το λιμάνι, άρα χάνονται πολλά χρήματα από τα εμπορικά πλοία τα οποία δεν αράζουν πλέον στο λιμάνι. Άρα έχουν περιοριστεί πολύ τα έσοδα τα εμπορικά. Και αυτό εν μέρη λόγω των ε, υψηλών ασφάλιστρων, τα οποία ζητούν οι ασφαλιστικές στην Ευρώπη. Άρα μία από τις αξιώσεις ε, της κυβέρνησης του Τσιμπουτή ήταν να περιοριστούν τα ασφάλιστρα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά της πειρατείας. Η συγκεκριμένη περιοχή από σήμερα θεωρείται ασφαλής. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια επιχειρηματολογία η οποία να δικαιολογεί την εκτόξευση των ασφάλιστρων. Γι' αυτό λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαμε να δράσουμε, να προσκαλέσουμε και εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιριών, εκπροσώπους και της κυβέρνησης του Τζιμπουτή, εδώ πέρα σε μια συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητηθεί ακριβώς το θέμα αυτό. Τέλος, Πρόεδρε. Το θέμα της λαθρέας αλίας στις ακτές της Σομαλίας. Και τα τοξικά απόβλητα τα οποία η Ευρώπη πετάει στις ακτές της Σομαλίας. Και εδώ η κυβέρνηση του Τζιμπουτή τόνισε ότι θα πρέπει να επιληθεί το ζήτημα αυτό και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς οικολογικής ασφάλειας. Άρα, παράλληλα με το πρόβλημα της πειρατείας, φαίνεται ότι ανακύπτουν δύο σημαντικά άλλα προβλήματα. Η παράνομη αλία και τα τοξικά απόβλητα. Αυτά από πλευράς μου και σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα τα οποία θα τα βρείτε και εκτενώς στην γραπτή έκθεση. Είμαι βέβαιος ότι η κυρία Νικολάη, η οποία κατέφτασε το μεταξύ και την καλωσορίζω, θα σας ε, διαφωτίσει και θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα. Oui, merci, Ευχαριστώ κύριε Παλεύσκη. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ελπίζω ότι θα είναι επικοδομητική η συζήτηση. Θα μιλήσω ρουμάνικα, διότι θέλω να είμαι σαφής και να μην χάσω τις αποχρώσεις διαφορές. Ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά πράγματα μετά από την παρουσίαση που έκανε ο συνάδελφος. Αυτές είναι οι... Αυτά είναι τα πορίσματα στα οποία κατέληξε η αποστολή μας. Θα ήθελα απλώς να πω ότι η επίσκεψη αυτή για μένα προσωπικά αλλά και για τον συνάδελφο ήταν ένα πραγματικό μάθημα. Ενημερωθήκαμε πάρα πολύ καλά για την πραγματικότητα, διότι πολλές φορές ο τύπος μεταφέρει λανθασμένες προφορίες που να αντιστοιχούν με τίποτα όταν βρίσκεται κανείς επί τόπου. Βέβαια διάρκεια αυτή τη επίσκεψη λοιπόν μπορέσαμε να σχηματίσουμε μια σωστή εικόνα της αποστολής Αταλάντα. Όσον αφορά το στρατιωτικό σκέλος αυτής της επιχείρησης, πιστεύω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ επιτυχή επιχείρηση του αλλά υπάρχει ένα μεγάλος κίνδυνος. Κατά την άποψή μου, η επιτυχία αυτής της αποστολής θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την μελλοντική κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και οι στρατιωτικές αρχές μας ανέφεραν διάφορους κινδύνους οι οποίοι απορρέουν από τα όρια της εντολής την οποία κινούνται, διότι πολλές φορές δεν μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά. Δίδω ένα παράδειγμα. ακόμη και αν μπορούν μέσω των εναερίων ε, περιπτώσεων να έχουν σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούν και τις μεθόδους, δεν μπορούν να παρέμβουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα να επηρεάσουν τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να διευκρινιστεί, να αναθεωρηθεί η εντολή. Επίσης, υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την εκεί περιοχή και μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία των ε, διαφόρων αποστολών. Μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι δεν μελετήσαμε ίσως πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις διαπραγματεύσεις για την αμοιβή που θέλουμε να δώσουμε έναντι προφορέ. Ίσως, λοιπόν, δεν μπορούμε να εκριζώσουμε αυτό το φαινόμενο της πειρατείας. Τέτοιου είδου έρευνες δεν μπορούν να τις κάνουν οι τοπικές αρχές. Διότι ίσως πρόκειται για οργανωμένα ε, δίκτυα εγκληματιών, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται, προέρχονται από την Ευρώπη, γι' αυτό ζητούν και αυτά τα υπέρον καλύτερα. Θα μπορούσε ίσως εδώ η Ευρωπόλ να κάνει μία πιο λεπτομερή και περιστατωμένη έρευνα για να μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε αυτά τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Ίσως θα μπορούσαν να έχουν και σχέση με άλλα τρομοκρατικά κινήματα και να χρηματοδοτούνται και από τέτοιου είδους δίκτυα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία εμπεριστατωμένη έρευνα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και την ε, ε, ειρήνη και την ασφάλεια σε εκείνη την περιοχή, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεδομένου ότι ακούγεται ότι υπάρχουν και διασυνδέσεις και σχέσεις με την ε, Αλκάιδα, Αυτό λοιπόν το θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο λεπτομεριακά. Επίσης θα ήθελα να γίνει η συζήτηση του θέματος των λύτρων που καταβάλλονται και με άλλους οι οποίοι ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα. Ε, και αναφέρομαι στα λίτρα που δίδονται για να απελευθερώνονται τα πλοία. Διότι αν δίδουμε τέτοιου είδους ποσά και δεν κάνουμε τίποτα άλλο, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να υποδαβλίζουμε περαιτέρω τέτοιου είδους ε, ε, πράξεις πειρατικές. Επίσης, Πιστεύω ότι το θέμα των δικαστικών ερευνών και των ποινικών κυρώσεων που θα επιβάλλονται για τέτοιου είδους ε, θέματα σε αυτούς οι οποίοι ή προστατεύουν ή αυτούς ε, οι οποίοι θέλουν ε, να δικάσουν τέτοιου είδους πειρατές θα πρέπει να εξεταστούν καλύτερα και να ενισχυθούν. Θα πρέπει το Λαντ και το Πούτλαντ να τα εξετάσουν περαιτέρω για να δούμε αν δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ερευνών που θα κάνουν οι υπεύθυνοι, αν δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα δίκτυο δικαστικών αρχών που θα ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα, ώστε να έχουμε πάντα τους κατάλληλους ε, δικαστές. Επίσης, ε, χώρους φυλάκισης. Δεν υπάρχουν πάντα οι κατάλληλες φυλακές για άτομα τα οποία διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις επιτόπου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα παρακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της κατάρτισης, της επιμόρφωσης για κάποιους αξιωματούχους και κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις. Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους δράσεις στην Ουγκάντα, αλλά δεδομένου ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να επιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Επίσης, ε, μου ανέφερε κάποιος ότι υπάρχουν ε, αξιωματούχοι οι οποίοι δεν έχουν ε, λάβει τις αμοιβέ τους εδώ και ένα χρόνο. Δεν μπορούμε λοιπόν να ενεργούμε αποτελεσματικά, να έχουμε άτομα επί τόπου, να ζητούμε να γίνεται και ε, συμμετοχή, να υπάρχει και συμμετοχή τους σε θαλάσσιες επιχειρήσεις και να μην τους παρέχουμε ένα σταθερό εισόδημα. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό το θέμα της χρηματοδότησης και των κονδυλίων που παρέχουμε, ε, καθώς και το θέμα της επιμόρφωσης των ε, ε, αστυνομικών αρχών, να το ξαναδούμε ώστε να μπορέσουμε να ενεργούμε αποτελεσματικά επιτόπου. Και θα ήθελα να κάνω και μια τελευταία παρατήρηση. Μας ζήτησαν να εμπλακούμε πιο αποτελεσματικά και πιο άμεσα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων οικονομικών προγραμμάτων επιτόπου για να δημιουργηθούν τα κατάλληλα έργα υποδομής, ε, κοινωνική ε, έργα υποδομής για να υποστηρίξουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και να καταπολεμήσουμε την υπερβολική ένδυα που είναι γενικευμένη. Εάν δεν ενεργήσουμε με πιο πρακτικό τρόπο, με πιο συντονισμένο τρόπο, κινδυνεύουμε ακόμη και αν είμαστε ένας από τους κύριους φορείς υποστήριξης της περιοχής και ξέρουμε ότι και στην Ιεμένη και στην Ουγκάντα η κατάσταση είναι πάρα πολύ λεπτή. Ίσως άλλες δυνάμεις διεθνείς θα μας υποκαταστήσουν, όπως η Κίνα Φερρυπίν, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γιατί πάρα πολύ ε, εμπεριστατωμένες αναφορές σας, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Πρώτα απ' όλα την επιτυχία αυτής της επιχείρησης και τον πιλωτικό της χαρακτήρα που είναι πρωταρχική σημασίας για να μπορέσει να αναπτυχθεί το στρατιωτικό ε, συντεταγμένη αυτή της ΚΕΠΑ. Το γεγονό ότι διαδραματίζει ε, ρόλο σημαντικό, ρόλο κινητήριας δύναμης Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση με την καταπολέμηση της πειρατεία είναι σημαντικό. Αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι οι εταίροι μα τρίτες χώρες, το ΝΑΤΟ, που λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο συνεργάτης, ο πιο κατάλληλα ε, οπλισμένος αν θέλετε για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και επίσης θα θέλαμε τον πολυσχεδή χαρακτήρα όλων αυτών των επιχειρήσεων να τον τονίσουμε. Έτσι μπορούμε να παρέμβουμε επί τόπου στη συγκεκριμένη περίπτωση Σομαλία, να, σε πολλούς τομείς, στον δικαστικό μεταξύ άλλων σε άλλους και μπορεί να αποτελέσει αυτό παράδειγμα το τι συμβαίνει στον κόλπο του Άντεν και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για όλη την περιοχή και του ειδικού και νου, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να εμπλακούν μπλακούν σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινο... πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις στρατηγικές, σε όλες τις ε, ε αποστολές που αφορούν την περιοχή αυτή της, ε, του κέρατος της Αφρικής, ιδιαίτερα στην περιοχή Σομαλίας. Πρέπει να σας πω ότι άρχισαν επαφές με εκπροσώπους της Somaliland. Θα πρέπει όμως περαιτέρω να τις ενισχύσουμε. αν ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, βεβαίως και το θέμα το ε, ακτοφυλακής της ασφάλειας και τάρτη των ακτοφυλάτων επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό. Θέλει κανένας να πάρει το λόγο. Ο κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Απλώς θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο ουσιαστικής ουσιαστική σημασία δίδουμε εμείς στην υποεπιτροπή μας στην ε, αποστολή Αταλάντα ευθύς εξ αρχής έχουμε προσδώσει η σημασία σε αυτή την επιχείρηση. Γιατί ιδιαίτερη. Πρώτα απ' όλα, διότι ήταν η πρώτη, είναι η πρώτη επιχείρηση θαλάσσης αέρος, στην οποία συμμετέχουν διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι είναι να γίνει κατά κάποιο τρόπο μια κοινή αποστολή όλης της ΚΕΠΑ. Έχει πιλωτικό χαρακτήρα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πρότυπο, μοντέλο, το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική κοινή πολιτική ασφάλειας. Δεύτερον, για τον ε, στόχο. Ποιο ήταν ο στόχος. Στην περίπτωση του κόλπου του Μπάνταν και στον ειδικό ωκεανό να εξασφαλίσουμε ασφαλείς θαλάσσιες με μεταφορές και διάβλους ασφαλείς για τη διέλευση των πλοίων. Έχουμε λοιπόν ένα νέο παράδειγμα της ελευθερίας διακίνησης από μια περιοχή του κόσμου στην άλλη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και μας εξήγησαν πώς αναπτύχθηκε αυτή η επίσκεψη. Θα ήθελα και εγώ να είμαι μέρος της ε, αποστολής σας, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα διότι ήμουνα στην Ισημερινό. Αλλά όπως γνωρίζετε, η χώρα μου προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιχείρηση αυτή Αταλάντα. Και τελικά θα ήθελα να αναφέρω και κάτι το οποίο είπε και η συνάδελφος και το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Δεν θα πρέπει μόνο να μπορούμε να ενεργούμε in του επί αλλά και στα κέντρα στα οποία ε, γίνεται και η πληρωμή των λίτρων. Ξέρουμε ότι στο ΣΥΤΙ, στο Λονδίνο, υπάρχουν ε, γραφεία δικηγόρων στα οποία γίνονται όλες αυτές ε, οι δοσοληψίες. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί για να έχουμε πάντα επιτυχείς επιχειρήσεις τέτοιου είδους. Ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Νικολάη, την συνάδελφο για τον απολογισμό της επίσκεψης. Θα μπορούσε να μας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες περί λαθραλίας για τους ισχυρισμούς επίσης περί απόρριψης τοξικών αποβλήτων Υπάρχουν βάσιμοι ισχυρισμοί κατά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάτι τέτοιο υπονοείται στην έκθεση. Είναι πράγματα όχι ευχάριστα, τα οποία θέλουμε να αποφεύγουμε, αλλά να το συζητήσουμε αν πράγματι υπάρχουν κατηγορίες ή κάποιοι τέτοιοι, τέτοιοι ισχυρισμοί. Να πω επίσης ότι δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιληθεί με στρατιωτικά μέσα. Αν και αποδέχομαι ότι πρόκειται περί μιας δοκιμαστικής πιλωτικής παρέμβασης και μπορεί να έχει πετύχει από στρατιωτικής απόψεως, όμως τις ρίζες του προβλήματος δεν τις αντιμετωπίζουμε. Στη Σομαλία και στην περιοχή εν γέννη. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και να δούμε το πρόβλημα με τους αρμοδίους στην περιοχή. Πρόκειται για έναν μηχανισμό τον οποίο ελέγχει η Αιθιοπία και που είναι μέρος ε, προβλήματος και τις λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να ρωτήσω, αν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήσατε και να ακούσατε κάποιες σκέψεις για την εμπλοκή του κλιμακίου εκπαίδευσης που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουγγάντα για μέλη των, για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Σομαλίας. Ε, δεν ξέρω τελικώ αυτοί ποιου θα υπηρετήσουν μετά από την κατάρτιση που παρέχουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σλίζακ. Ε, εγώ από την πλευρά μου Ο συνάδελφος είπε ότι έχουμε καλή συνεργασία, υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Όμως, από ό,τι ξέρουμε, στην περιοχή υπάρχουν και σκάφη τρίτων χωρών με παρόμοιους στόχους. Ρωσικά και κινέζικα συγκεκριμένα. Το σχολιάσετε καθόλου αυτό με τους εκπροσώπους της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Υφίσταται κάποια συνεργασία ή τουλάχιστον συντονισμός με τα σκάφη των τρίτων χωρών. Πρόσφατα, ένα ρωσικό πολεμικό σκάφος έλεπε δράση που γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα. Θυμάστε την εξαφάνιση των πειρατών και όλοι θαυμάσαμε τους Ρώσους για την αποτελεσματικότητά του, αλλά δεν ξέρω αν κινούνται με βάση του ίδιου ε, κανόνες που ακολουθούν τα δικά μας θέματα. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία μεταξύ Ρώσων και ημών. Ήταν. Ευχαριστώ. σα ευχαριστώ. Κύριε Νικολάη. Για να απαντήσω, δεν είναι κύριε Γκόμες. Αγαπητοί συνάδελφε, οι ισχυρισμοί περί λαθραλίας από σκάφη τρίτων χωρών. Ε, τι να σου πω, δεν έχω δει αποδείξεις. Δεν γνωρίζω. Για την απόρριψη τοξικών αποβλήτων, οι αρχές του Τζιμπουτή διατύπωσαν αυτές τις κατηγορίες. Μίλησαμε με τον Υπουργό Μεταφορών, αλλά και με τον Πρόεδρο της ε, Βουλής ε, και ο κ. Σελέτσικη θα το επιβεβαιώσει αυτό το οποίο λέω, ε, οι ισχυρισμοί αυτοί ακούστηκαν κατά τη διάρκεια εκείνη τη ε, συζήτησης. Και θα είμαι πολύ προσεκτική, δεν υπάρχουν αποδείξεις περί αυτού. Καταγράψαμε τους ισχυρισμού, τις κατηγορίες αν θέλετε, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι πράγματα που αξίζει το κόπο να συζητήσουμε εδώ. Όσον αφορά τώρα την Ουγγάντα να σας ενημερώσω ότι το κλιμάκιο έχει αποτελεσματικότητα, εκπαιδεύει στρατιωτικούς. Τώρα από εκεί πέρα αυτές οι δυνατότητες και αυτά τα στελέχη τι θα κάνουν, έχω τις εμβολίες μου. Από νομικής απόψεως, τα στελέχη που εκπαιδεύσαμε πρέπει να αξιοποιηθούν από την Σομαλία. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι η Σομαλική κυβέρνηση είναι μεταβατική κυβέρνηση. Συνεπώς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος με την συνήθεια ευρωπαϊκή έννοια του όρου. Θα χρειαστεί πολύ χρόνος για να δράσει η Σομαλία ως, ε, αν θέλετε, ευρωπαϊκό κράτος από απόψεως αποτελεσματικότητας. Μετά λοιπόν την ε, εκπαίδευση ε, και εκπαιδεύσουμε και στρατιώτες και αστυνομικού. Πιστεύω ότι η εμπλοκή της ε, Σομαλίας θα είναι πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Αυτή είναι η θέση μου προς το παρόν. Τώρα, όσον αφορά την συνεργασία με τις άλλες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ο Γάλλος επικεφαλής μας είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο ότι υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο. Διευκρίνησε όμως ότι οι εντολές των κατέρωθων δυνάμεων είναι διαφορετικές. Εμείς έχουμε την Αταλάντα, μια δομημένη επιχείρηση. Το ΝΑΤΟ, που έχει επίσης παρουσία στην περιοχή αντίστοιχα, οι Αμερικανοί λίγο πάντως ασχολούνται με την ε, πειρατεία. Φυσικά θέλουν να ασκούν επιρροή στην περιοχή, αλλά κατά την απόψή μου έχουν τα μάτια περισσότερο στραμμένα στην Αραβική Χερσόνησο, προς την Ιεμένη και λιγότερο προς το Σουδάν. Τους Αμερικανούς, εν πάση περιπτώσει, όπω είπα, του απασχολεί λιγότερο η πειρατεία. Προσπαθούν να οικοδομήσουν ε, σχέσεις με τι τοπικέ αρχέ, μέσω μικρών έργων για οικονομική ανάπτυξη, για σταθερότητα, κοινωνικές παρεμβάσεις κλπ. Ό,τι άλλο συμβαίνει στην περιοχή, πάντως αφορά τα ίδια τα κράτη μέλη, πρόκειται για εθνικέ δράσει. Γι' αυτό ξαναλέω ότι η Αταλάντα είναι μια διαφορετική υπόθεση. Πάντω συνεργαζόμαστε, ανταλλάσσουμε πληροφορίε και όταν πρόκειται για κοινέ ε, ενέργειε φυσικά, αυτό είναι αυτονόητο. Έχουμε μετά εκτός από τους Κινέζους και την Ιαπωνία, η οποία προσπαθεί να ιδρύσει μια στρατηγική βάση στον Τζιμπουτί και υπάρχει και η Ρωσία. Είναι κράτη τα οποία προσπαθούν να προστατεύσουν τις εμπορικές ανταλλαγές τους με πολεμικά σκάφη τα οποία περιπολούν στην περιοχή, στον Τζιμπουτί και στον Ινδικό ωκεανό. Όσον αφορά τώρα το πλοίο που κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις, πρόκειται για ειδήσει που ήταν στα πρωτοσέλιδα. Εκεί δεν ε, έχουμε αρκετέ πληροφορίε. δεν πήραμε από του συναδέλφου μα αρκετέ πληροφορίε για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα. Όπω είπα αυτά και το γνωρίζετε, ήταν στα πρωτοσέλιδα. Όλοι άκουσαν ε, φήμε περί του επεισοδίου. Κανεί όμω δεν έχει σαφή εικόνα, διότι δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε και συνεπώ δεν μπορούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα. Κύριο Ζαλεύσκη. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Λίσεκ, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Νικολάη το εξής. Επανελειμμένα έχουν γίνει συναντήσεις των συντονιστών της επιχείρησης Αταλάντα και των στρατευμάτων, των επικεφαλής του ΝΑΤΟ και των Αμερικανικών στρατευμάτων. Και οι δραστηριότητε αυτές είναι σε εξέλιξη, όπως είπε και η κυρία Νικολάη και τα άλλα σκάφη τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή κινέζικης και ρωσικής προέλευσης κυρίως, ε, δρούν κατά, κατά εθνικών, σύμφωνα με εθνικές εντολές και δεν είναι τμήμα των επιχειρήσεων κατά της πειρατείας. Φυσικά τα σκάφη αυτά αναλαμβάνουν δράση μόνον όταν απειλούνται τα σκάφη σημαίας τους. Και τα δικά τους λοιπόν πρότυπα ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές, γιατί μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση, την περίπτωση της Ρωσίας. Φυσικά τα πρότυπα που χρησιμοποιούν διαφέρουν από εκείνα τα οποία εφαρμόζουν τα σκάφη ευρωπαϊκής ή αμερικανικής σημαίας. Ή, εν πάση περιπτώσει, τα σκάφη τα νατοϊκά. Ανεξάρτητα από το τι συνέβη στους πειρατές οι οποίοι απήγαν ε, ρωσικό σκάφος, πρέπει να πω ότι δεν ε, εξαφανίστηκαν πολύ απλά χωρίς να έχει υπάρξει δικαστική απόφαση. Δεν έχω οποιαδήποτε πληροφορία και φυσικά αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ανησυχεί ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά σκάφη, γιατί η καταπολέμηση της πειρατείας θέλουμε να γίνει με πλήρη σεβασμό του δικαίου. Και οι στρατιώτες οι οποίοι συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελλάδα συλλέγουν αποδεκτικά στοιχεία για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία σε ό,τι αφορά τα άτομα που κατηγορούνται για πειρατεία. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσοι κατηγορούνται για πειρατεία είναι όντως πειρατές σε ό,τι αφορά τώρα τις ρωσικές ε, δράσεις. Η ρωσική δράση καταδεικνύει ότι τα πρότυπα τα οποία εφαρμόζουν οι Ρώσοι εταίροι είναι πολύ απλά διαφορετικά. Ευχαριστώ. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Σκίνερ ζήτησε το λόγο. Χαίρομαι, διότι είδα σε ένα κατάλληλο ότι θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Όπως λέει εδώ, να, κάτι, να κάνει για να απαγορεύσει την καταβολή αυτών των λίτρων. ήταν, όπως είπε και ο συνάδελφος, τρεις χώρες. Ίσως η χώρες, οι κυρίες, δύο-τρεις χώρες οι οποίες κάνουν και τις μεγάλες τα ασφάλειες οι οποίες θα μπορούσαν να δουν. Και ξέρουμε βεβαίως τι ζητούν οι διάφοροι. Όταν θα μπορέσουμε λοιπόν να γνωρίζουν όλοι τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να κάνουν ίσως, θα μπορούσαμε από κοινού με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και άλλους να το όλο θέμα. Δεύτερον, το θέμα αυτό διαφορετικό από την καταβολή ε, λίτρων ατομικά για κάποιον. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, φορές ε, ε, καταγραφή τέτοιου είδους γεγονότων εκ μέρους μιας οικογένειας ενός ατόμου. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε για τις κυβερνήσεις και μεταξύ των κυβερνήσεων της Ευρώπης ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν είτε και ποιοι όχι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να γνωρίζουμε σωστά ποιοι ναι και ποιοι όχι θέλω κάνει τέτοιο. Θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να μας να προσθέσουν κάτι για το γεγονός ότι η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας κάνει χώρο για 20 χιλιάδες άτομα τα οποία θα πρέπει να είναι επιτόπου. Ποτέ όμως νομίζω ότι δεν ξεπεράστηκαν οι 8.000. Αυτό είναι κάτι που το αναφέρατε στις συζητήσεις σας. Η ΙΓΚΑΤ προτείνει να αλλάξουν οι κανόνες που ισχύουν ώστε να μπορέσουν να καταπολεμήσουν απευθείας την Ασαμπάπ ε, και να μπορέσει τα, τα Ηνωμένα Έθνη να είναι υπεύθυνα για τέτοιου είδους αποστολές. Μπορείτε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται. Πάρα πολύ ε, σύντομα λέει ο Πρόεδρος γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο που είχαμε για τη Σομαλία και θα πρέπει να συζητήσουμε και ένα εξίσου σημαντικό θέμα μετά. Τα θέματα των Παλαιστινιακών εδαφών το θέμα το συζητήσαμε και η πολύ ειλικρινής και απλή απόφαση είναι ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια των ατόμων τα οποία χρησιμοποιούν εκεί. Αλλά Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτέ τι αποστολέ, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι τα πράγματα βαίνουν καλώ. Απλώ και εγώ θέλω να συμφωνήσω με την κυρία Νικολάη, ο πρόεδρο. Λυπούμε που δεν μπόρεσαν περισσότερα άτομα να λάβουν μέρο στην αποστολή αυτή. Όπω ξέρετε, έχουμε αυτό το παράλογο σύστημα των ποσοστώσεων και για τις ε, αποστολές 10 άτομα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι είναι παράλογο και νομίζω ότι εξορισμού οι αποστολές οι δικές μας, τις δικές μας επιτροπή του ή άλλως λαμβάνουν χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω όμως ότι όταν πρόκειται για τόσο σημαντικά θέματα, τόσο σημαντικές και επιτυχείς αποστολές, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία συζητούμε και μεταξύ μας και με άλλου συναδέλφους. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μαζί μας είναι ο κύριος Κλάμπενάουερ, διοικητή μη στρατιωτικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνταγματάρχη Αλάνθος Γάς, αρχηγό της αποστολής Ομπαμ Γαφά και τον αρμοστή Χένρικ Μάλκφουις, αρχηγό της αποστολης Ιου Πολ Corps. Πρόκειται για αποστολές στα παλαιστινιακά εδάφη που δυστυχώς, δυστυχώς απεικονίζουν πάρα πολύ καλά την ε, εικόνα για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειρηνευτικές Δυνάμεις στα Παλαιστινιακά εδάφη. Είναι απαραίτητες τέτοιου είδους ε, αποστολές και είμαστε, πρέπει να πω, και πολύ ε, μετριοπαθείς αυτές τις αποστολές. Πρόκειται για αποστολές από το 2005-2006 η Ούμπα Μραφά αναπτύσσεται, αναπτύχθηκε μετά από την μονομερή αποχώρηση του Ισραήλ από την Γάζα στην περιοχή της Ράφα, αλλά συνέχισε να επιχειρεί διότι έφτασε εκεί η Χαμάς και η Ιούπολ Κόψ άρχισε το 2006 στην ε, Δυτική Λωρίδα συνεργάζεται για την ε, επιμόρφωση των ε, τοπικών αστυνομικών δυνάμεων. Επίσης, όπως ξέρετε, αναθεωρείται τώρα η όλη πολιτική μας για τα Παλαιστινιακά εδάφη. Όπως θέλει και λέει θα έπρεπε να έχουμε μια ευρύτερη ε, πολιτική. Είναι Επίκαιρο λοιπόν αυτό το θέμα της αναθεώρησης των αποστολών αυτών. Είναι λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρον το όλο θέμα και ευχαριστώ τους δύο επικεφαλείς των αποστολών που είναι σήμερα μαζί μας και την γραμματεία του Συμβουλίου που μας βοήθησε. Ο κύριος Κλόπενχάουερ, ο συνήθως, ως διοικητής αυτής της μη στρατιωτικής επιχείρησης, είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Παρακαλώ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σα και θα ήθελα καταρχά να σα ενημερώσω ότι χαίρομαι για την, ε, το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τις ε, επιχειρήσεις μας και επίσης χαίρομαι για το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την αποστολή στην Παλαιστίνη και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα για να συζητήσουμε τις ε, αποστολές της ΚΕΠΑ Ακούσατε του επικεφαλής των αποστολών στην Αφγανιστάν, στο Κωσυφοπέδιο, στη Βοσνία, Αρζεγοβίνη και στη Γεωργία. Και να συμπληρώσουμε λοιπόν την εικόνα σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για τις αποστολές μας στην Μέση Ανατολή. Θα ακούσουμε μετά και τους υπόλοιπους, ε, τους ταγματάρχη Φαγκουέρες και τον Αμμουστή Όπως είπε ο πρόεδρος σας, Έχουμε δύο αποστολές στην περιοχή από τα τέλη του 2005 αρχές του 2006 και μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές οι αποστολές αυτές, αλλά επιτελούν το στόχο το πολιτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υποστήριξη της ειρήνευσης και την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών. Ένα ασφαλές κράτος ε, του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός. Η ειρηνευτική μας ε, αποστολή στην περιοχή είναι βασικά συμβουλευτική φύσεως και συμβάλλει στην ασφάλεια και στο κράτος δικαίου στη Δυτική Όχθη και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, το τονίζω αυτό, ότι συμβάλλουμε δηλαδή στην ασφάλεια και στο κράτος δικαίου στη Δυτική Όχθη σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση δυνατοτήτων ε, των Ισραηλινών ε, και Παλαιστινιακών δυνάμεων. Θα αφήσω στον ε, κύριο Μόλκβεστ να, παρουσιάσει τις πτυχές της αποστολής αυτής σε ό,τι αφορά ε, το σύστημα των... της φύλαξης των συνόρων μεταξύ της κυβέρνησης ε, της Παλαιστίνης και της κυβέρνησης ε, του Ισραήλ και της αρχής της Παλαιστίνης ε, έγινε μια τέτοια συμφωνία στις αρχές του 2006 η οποία αποτελεί τη βάση για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφώνησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εποπτεύσει τις δραστηριότητε στην περιοχή. Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρός σας από τότε που ανέλαβε η Χαμά στη Γάζα ανεστάλλει από τις αρχές του 2007 η αποστολή αυτή Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε όταν το επιτρέψει η πολιτική κατάσταση. Και ο κύριος Φοζράς, ο συνταγματάρχης Φοζράς θα σας δώσει τις σχετικές πληροφορίες. Θα γνωρίζετε ίσως ότι συμμετέχουν και άλλες χώρες στην περιοχή. Έχουμε πολλαπλές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διμερείς ε, ε, ενέργειες από τα κράτη-μέλη και COPS έχει συντονιστικό ρόλο για την διοχέτευση βοήθειας προς την ε, Παλαιστινιακή πολιτική αστυνομία. Θα πρέπει να πω ότι οι αποστολές οι οποίες ε, αναπτύσσονται λειτουργούν σε ένα πολύ περίπλοκο πολιτικό περιβάλλον και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. ο ύπατος αρμοστής εξακολουθεί να ανησυχεί πάρα πολύ για την κατάσταση στη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι είναι πρόθυμη τον προηγούμενο Ιούνιο να συνεχίσει για να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για την ε, αναδιάρθρωση της οικονομίας της παρακολουθούμε στενά τις ε, ευρωπαϊκές ε, δράσεις για να αρθεί αυτό το αδιέξοδο στη Γάζα. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα δώσω το λόγο στον Συνταγματάρχη. Σας ευχαριστώ. Η ήταν η πρώτη αποστολή, 2005. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Φωσράση για να μας παρουσιάσει τα σχετικά. Merci, Monsieur le Président. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο αλλα Αλά Φοζεράς της Γαλλικής Χωροφυλακής στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως επικεφαλής της ΕΟΜΠΑΜ. Η ΕΟΜΠΑΜ είναι μια δύναμη σε ετοιμότητα, να το διευκρινίσω αυτό από την αρχή. μια εφεδρεία η οποία θα αναπτυχθεί με το που θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θέλω να θυμίσω τους αρχικούς λόγους της παρουσίας μας στην περιοχή και θα σας περιγράψω και την σημερινή κατάσταση. Τον Αύγουστο του 2005 ο Ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε από την λωρίδα της Γάζας και διέλυσε τους ε, εβραϊκούς οικισμούς της περιοχής. Η περιοχή λοιπόν πέρασε στα χέρια της ε, Παλαιστινιακής Αρχής. Τον, τον ε, έλεγχο όμως της ενεργής καθώς και των χωρικών υδάτων της περιοχής καθώς και τον έλεγχο των συνόρων μεταξύ Γάζας και Ισραήλ τον διατηρεί το Ισραήλ. Από τότε του Ισραήλ ελέγχει όλες τις κινήσεις ε, προσώπων και εμπορευμάτων ε, που εισέρχονται ή εξέρχονται από την λωρίδα της Γάζας. Υπό τις νέες συνθήκες και υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και χάρη στη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ οι Ισραηλοί και οι Παλαιστίνοι συμφώνησαν για τις συνθήκες πρόσβασης στην περιοχή. Στόχος αυτής της συμφωνίας, όπως γνωρίζετε, ήταν η ρύθμιση της εισόδου και εξόδου των Παλαιστινίων από και προς το Ισραήλ. Από και προς λοιπόν την λωρίδα της Γάζας αλλά και μεταξύ της λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης. Η συμφωνία προβλέπει την δημιουργία σημείων διέλευσης για τα εμπορεύματα, για τους σκοπούς των εξαγωγών ε, συγκεκριμένα έχουμε το πέρασμα Σολκάρνη. Ε, έχουμε όμως μετακινήσεις και εντός της λωρίδας ε, της Γάζας και προβλέπεται και δημιουργία αεροδρομίου και λιμανιού. Τώρα, όσον αφορά την Ράφα, η Ράφα βρίσκεται στον νότο, στα σύνορα δηλαδή της λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Οι Ισραηλινοί η Παλαιστίνη, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δύο άλλα μέλη του κουαρτέρου, δηλαδή τα Ηνωμένα Εθνική Ρωσία, όλα λοιπόν τα εμπλεκόμενα μέρη, συνειδητοποίησαν ότι το πέρασμα της ράφα αποτελεί ειδικό θέμα και ότι πρέπει να αναζητηθεί, να εξευρεθεί ειδική λύση. Το σημείο αυτό είναι υπό Παλαιστινιακό έλεγχο. Το παρακολουθεί όμως τρίτη ανεξάρτητη αρχή για να, για να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα διεθνή πρότυπα. Παλαιστινοί και Ισραηλινοί κάλεσαν επισήμω την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ακριβώ αυτόν τον ρόλο τη επιτήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε την πρόσκληση και η Ιούμπαμ Ράφα προ το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στην περιοχή με τη μορφή κλιμακίου αστυνομική δύναμη. Πρόκειται, αν θέλετε, για κλιμάκιο υποστηρικτικό του ελέγχου των συνόρων ιδρύθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 2005 συγκεκριμένα. Η εντολή μας συνοψίζεται στην ενεργό επιτήρηση, επαλήθευση της δυνατότητας των Παλαιστινιακών αρχών να επιτηρεί τα σύνορα με ασκεί αστυνομικά καθήκοντα καθώς και τελωνιακούς ελέγχους. Οι βασικές αρχές σύστανται στην ε, διασφάλιση της κανονικής κυκλοφορίας Παλαιστινίων μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας, λαμβανωμένων υπόψη των αναγκών ασφαλείας. Η χρήση του σημείου διέλευσης στη Ράφα εξυπηρετεί φυσικά τους Παλαιστινίους αλλά και διπλωμάτες, επενδυτές, εκπροσώπους ε, ανθρωπιστικών οργανώσεων ε, ή άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών. Το συνολικό φυλάκιο της Ράφα χρησιμοποιείται επίση και για την εξαγωγή προϊόντων μέσω Αιγύπτου ή προς την Αίγυπτο αν θέλετε. Για να σας δώσω μια γενική εικόνα, το φυλάκιο ελέγχει διαβατήρια, ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, όπως σε κάθε άλλο συνοριακό φυλάκιο. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για Παλαιστινιακό έλεγχο υπό την επιτήρηση όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καθιάσουν και τους ε, Ισραηλινούς δημιουργήθηκε άλλο ένα σενεργό φυλάκιο προς το Ισραήλ το οποίο στελεχώνεται από Παλαιστινίους όσο και Ισραηλινούς τελωνιακούς με επιτήρηση με ανεξάρτητη επιτήρηση και εκεί. Στα δύο αυτά σημεία η UBM, λοιπόν ασκεί τον ρόλο του τρίτου ενεξάρτητου παρατηρητή και συμβάλλει στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνη. Ω ουδέτερο τρίτο μέρο παρεμβαίνουμε και υποβοηθούμε τι διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο αμέσω εμπλεκομένων για την αναζήτηση λύσεων. Η UBM ξεκίνησε όπω είπαμε 25 Νοεμβρίου του 2005 έως τι 25 Ιουνίου του 2006 σε πρώτη φάση Χάρη στην αποστολή αυτή, 280.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα καθη... καθημερινά. Χίλιοι άνθρωποι την ημέρα τουλάχιστον. Το άνοιγμα του φυλακίου της Ράφα είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την Λωρίδα της Γάζας που αφορά την πρόσβαση στην περιοχή. Εάν πετύχαινε το πρώτο σκέλος της προσπάθειας, αυτό θα άνοιγε τον δρόμο και για το αεροδρόμιο καθώς και για το λιμάνι. Η στη Ράφα διαδραμάτισε πολιτικό ρόλο κλειδί, δεδομένου ότι πρόκειται για το μόνο συνεργό φυλάκιο στα σύνορα Αιγύπτου Λωρίδες της Γάζας. Το 2005 λοιπόν ως το 2006 Παλαιστίνοι επιτέθηκαν σε Ιρανιές δυνάμεις και εισέλαβαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη, τον ε, Τζιλάντ Σαλίτ. Εμείς προσπαθήσαμε να απαγορεύσουμε την εκτόξευση ροκετών Κασάμ και από το 2007 το φυλάκιο ανοίγει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος. Από τις 10 Ιουνίου μετά του 2007 μέχρι σήμερα έχουν ανασταλεί οι επιχειρήσει μα. Τον Ιούνιο του 2007, όπω γνωρίζετε, η Χαμά ανέλαβε τον έλεγχο τη Λωρίδα τη Γάζα. Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει απευθεία επαφές με την Χαμάς και το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φυλάκιο λοιπόν στη Ραφά έκλεισε και νομικά τουλάχιστον δεν υφίσταται έκτοτε, δεν έχει λειτουργήσει δηλαδή. Νομικά εννοώ με βάση τουλάχιστον τη συμφωνία του 2005. Παρ' όλα αυτά, το κλιμάκιο της UBAM στη Ράφα έχει την ε, σημασία που είχε διότι όπω είπα διευκόλυνε συνολικά τη διέλευση άνω των 430.000 ανθρώπων ως ε, το 2007 συγκεκριμένα. Συνεχίζει να αποτελεί το πέρασμα λωρίδα επικοινωνία ζωτική σημασία για την λωρίδα της Γάζας από τότε που τον έλεγχο ανέλαβε το 2006 η Χαμάς. Η περιοχή βρίσκεται σε κρίση από ανθρωπιστικής απόψεως. Αντιμετωπίζονται συνεχώς ε, στρατιωτικές εισβολές των Ισραηλινών, ε, συν οι ε, διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων, αντιμαχωμένων παρατάξεων των Παλαιστινίων. Αυτή τη στιγμή είμαστε ε, έτοιμοι να αναπτυχθούμε πλήρως σε τρεις εβδομάδες. Είμαστε σε επαφή με τις εμπλεκομένες πλευρές και με τους άλλους εμπλεκομένους φορείς στην περιοχή. Ο σκοπός είναι να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας στην περιοχή. Η Γιούμπαμ συνεχίζει να ε, υποβοηθά σε θέματα τριωνιακών και αστυνομικών ελέγχων. Είμαστε παρόντες, δίνουμε διαλέξεις, συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας, συμμετέχουμε σε σχεδιασμό και προγραμματισμό και επίσης συλλέγουμε πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή. Εν για τα δύο χρόνια που είμαι στην περιοχή, θα έλεγα ότι τον Δεκέμβριο, 8 Ιανουάριου του 9 είχαμε σημαντικά επεισόδια και βεβαίω έχουμε και το επεισόδιο, τα επεισόδια του Ιανουαρίου του 2010, γνωστό στο Λίσκο, που προσπάθησε να προσεγγίσει τη Γάζα, κάτι το οποίο αποδεικνύει την ε, ανάγκη ύπαρξης της στην περιοχή, καθώς και την προσθέμενη αξία που μπορεί να συνεισφέρει. Η UBAM υπήρξε ένα πολύτιμο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια της να συμβάλλει στην ειρήνευση στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ah, euh, Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο γνωστής Henrik Μακουίστ, αρχηγός υποστολής Γιούπολ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με καλέσαν ε, στην υποεπιτροπή σας σήμερα και μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ενημερώσω για την αποστολή μας UPOL COPS. Πρόκειται για μια αποστολή που άρχισε ως διμερής ε, αποστολή υποστήριξη αστυνομία Ευρωπαϊκή ε, της ε, ε, Ηνωμένου Βασιλείου έγινε από το 2006 και μετά διεθνή. Έχουμε μέλη, 23 μέλη από 17 κράτη-μέλη και συμμετέχουν τέχουν προς το παρόν από τρίτες χώρες, Καναδί και αργότερα ίσως θα έχουμε καινούριους. Προς το παρόν μόνο από τρίτες χώρες, μόνο έχουμε Καναδούς. Είμαι υπεύθυνο αυτής της αποστολής από την αρχή του παρόντος έτους. Είμαι ο Χένρικ Μάλκμιστ. Ποια είναι η αποστολή μας. Να κάνουμε διάφορες ε, ε, ε, ρυθμίσεις και βοηδεστικέ ε, ρυσίες στα πλαίσια της παρακολούθησης, να κάνουμε την μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, να ασχοληθούμε με θέματα ποινικού δικαίου. Ασχολούμεθα μέχρι το 2008 μόνο με αστυνομικές επιχειρήσεις. Τώρα μας έχουμε και ένα δεύτερο πυλώνα που είναι αυτός Τη παρακολούθηση όλων των θεμάτων του κράτους δικαίου. Δεν ασχολούμεθα λοιπόν μόνο με θέματα που αφορούν τα αστυνομία αμυγό. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε πολύ προσεκτικά, διότι όλα εξαρτώνται από τους Παλαιστινίους και ζητούνται από τους Παλαιστινίους. Βεβαίως, εργαζόμαστε σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς προδιαγραφές και κανόνες και συνεργαζόμαστε και με τα ε, γραφεία της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα γραφείο χρηματοδότηση το οποίο υπάρχει στην Ιερουσαλήμ και εμείς ε, καταρχήν ως τέτοιου είδους αποστολή δεν έχουμε μεγάλη χρηματοδότηση, μόνο χρηματοδοτούμε μικρά προγράμματα, αλλά δίδουμε συμβουλές σε θέματα αστυνομίας και κράτου δικαίωση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι συντονίζουμε τις δραστηριότητες μας και με τις άλλες παρούσες ε, διεθνείς αρχές που είναι εκεί. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί διεθνείς προγραμματές είναι παρόντες. Πρόκειται για ενδιαφέρουσες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την εντολή μας, εμείς αυτό το που κάνουμε είναι να υποβοηθούμε τη μη στρατιωτική αστυνομία της Παλαιστίνης PCP για την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης της αστυνομίας. Και σύμφωνα με την εντολή μας επίσης προσπαθούμε να παρέχουμε συμβουλές και να ε, παρακολουθούμε τις δραστηριότητες της μη στρατιωτικής αστυνομίας. Δεν ε, κάνουμε εποπτεία των ε, και έλεγχο. Το μόνο το οποίο κάνουμε λοιπόν να παρέχουμε συμβουλές και όπως σας είπα ε, σε θέματα που αφορούν και το ποινικό δίκαιο. Και επίσης πρέπει να πω ότι συντονίζουμε και διευκολύνουμε τα σχέδια από κοινού άλλων φορέων. Εδώ θα ήθελα να σας πω πώς έχει παρούσα κατάσταση στα πλαίσια της αποστολής μας. Θα σας μιλήσω για τις τερικές διαδικασίες και τις σχέσεις και την ε, προκλήσεις μας. Πώς έχουν τα πράγματα. Όπως σας είπα, έχουμε δύο κυρίους πυλώνες δραστηριότητες. Θα σας μιλήσω για τον πρώτο, που είναι παροχή συμβουλών στον τομέα της αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε, ε, ασχολούμεθα με τέσσερις τομείς επιχείρησης. Πρώτα απ' όλα με την ε, μπλε αστυνομία, με την περιπολίες, με θέματα ε, που ασχολούνται οι detectives, με έρευνες. Τρίτος τομέας αξιοπιστία, εποπτεία. Προσπαθούμε να δώσουμε λοιπόν συμβουλές στην PCP για να μπορέσει να έχει αξιόπιστους σύγχρονους μηχανισμούς λειτουργίας. Τέταρτος τομέας, ε, υποστήριξη και επιμελητή. δεύτερος πυλώνας τώρα, ο τομέας του κράτους δικαίου. Εδώ Έχουμε εμπειρογνώμες σε θέματα φυλακής, εισαγγελείς, ε, δικηγόρους, νομικούς, πρώτα απ' όλα σε θέματα ε, δικαστηρίων, ρευνών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, ε, φυλακές και νομική προστασία. Εδώ τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Πρέπει να σας πω ότι η αστυνομία, όπως ξέρετε, ενεργεί ε, αν θέλετε, από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα σε αυτό το τομέα. Και αυτό γίνεται και στην Παλαιστίνη. Εδώ ε, βλέπετε κάποιους τομείς στους οποίους παρεμβαίνουμε. συμμετείχαμε στην ε, υπογραφή μνημονίου μεταξύ των γελικών οργών και της μη στρατιωτικής αστυνομίας. Και εδώ αναφέρονται οι τομείς συνεργασίας μεταξύ αυτών των δύο θεσμικών φορέων, διότι στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή πώς εργάζεται κανείς όταν έχει να κάνει έρευνα, όταν υπάρχει ε, εγκληματική ενέργεια, πώς ε, ε, αναθέτουν οι ανακριτικές αργές κάποια καθήκοντα σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να κάνουν έρευνα κτλ. Επίσης, τους τελευταίους 6 με 8 μήνες παρήχαμε τεχνική βοήθεια για το νέο ποινικό δίκαιο Και αυτό ήταν μέρος της αποστολής μας, κυρίως πώς θα βελτιωθεί ο τομέας των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Και θα υπάρχει στο μέλλον προεδρικό διάταγμα για να μπορέσουν να κατοχυρωθούν αυτά τα δικαιώματα. Επίσης, κάνουμε ειδικά μαθήματα επιμόρφωσης στον τομέα της εγκληματολογίας και της ε, καταπολέμησης διαφθοράς για δικαστές, μεταξύ άλλων, και τελικά επισκόπηση ε, του όλου συστήματος ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, τα αφορούν ισότητα των φύλων. Είναι θέματα με τα οποία ασχολούμεθα εγκαρσίως, δηλαδή για όλες τις δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσουμε. Πού ακριβώς είμαστε. Στο τμήμα ανάπτυξης στρατηγικής της αστυνομίας, στο Υπουργείο Άμυνα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο κέντρο επιμόρφωσης της ε, ε πολιτικής, στρατιωτικής ακαδημίας της Ιεριχούς που θα αρχίσει να λειτουργεί από του χρόνου το Μάιο. Προσπαθήσαμε επίσης εφέτος να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα που αφορούν τη δική μα εσωτερική διαδικασία. Δεν θέλω να σα κουράσω με τέτοιου θέματα, απλώ το αναφέρω για να μπορέσουμε να πούμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε σωστά και αποτελεσματικά ε, αποτελέσματα θα πρέπει να έχουμε και τον σωστό τρόπο εσωτερικής μας διοίκησης. Γι' αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε καλύτερα το όλο σύστημα και κυρίως τα θέματα συνεργασίας των διαφορών τμήματων να το βελτιώσουμε. Σε όλα τα φάσματα των δραστηριοτήτων μας. Εδώ βλέπετε με ποιους φορείς πρέπει να έχουμε σχέσεις στα πλαίσια της εντολής μας. Ε, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή ε, ε Είπα για τα θέματα κατάρτισης NNGF ε, Και δεδομένου ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που καταρτίζουν τις ε, αστυνομικές αρχές πράσινη ασφάλεια, όπω λέγεται, πρέπει να συνεργαζόμαστε και με του. Επίση, με τα διάφορα υπουργεία στην Παλαιστίνη, εκτό από αυτά του Ισραήλ, με τον ε, Γενική Εισαγγελία, με τα δικαστήρια και με την PCP. Και πρέπει να σας πω ότι σε εβδομαδιαία βάση εγώ συναντώ τον υπεύθυνο της ε, αστυνομίας, της στρατιωτικής αστυνομίας. Επίσης έχουμε σχέσεις και με τον ε, υπεύθυνο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι μελλοντικές προκλήσεις μας σε... αναφορά αφορά τις δραστηριότητές μας, διαδικασία ειρήνευσης, χρειάζεται να υπάρξει πρόεδρος για να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε το Παλαιστινιακό Σύστημα Ασφαλείας. Αυτό ακούγεται και σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Θα πρέπει κάπου να δει κανείς το φως στο τέλος του τούνελ για να νομιμοποιήσει τις δράσεις τις οποίες αναλαμβάνει. Και αυτό είναι κίτρινο. Κάτι άλλο είναι για το μέλλον που μας απασχολεί είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την υπεροχή την αστυνομία της Παλαιστίνης σε σχέση με τους άλλους παρεμφερείς φορείς που δραστηριούνται επί τόπου. Επίσης, σας είπα επίσης ότι όλο το θέμα ε, του ε, δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συνεργαστούμε. Τώρα, από εσωτερικής πλευράς. Τι θέλουμε να κάνουμε και αυτούς τους νέους στρατηγικούς μας στόχους να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην συνεκτικότητα των αποστολών και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δωρητών. Ε, ο συντονισμός των, ε, των δραστηριοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ε... Επίσης, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται για μας. Η αύξησή μας βεβαίως είναι κάτι που εξαρτάται από εδώ και βεβαίως έχουμε, ε, γι' αυτό έρθει σε διαπραγματεύσεις και με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Τα θέματα των σημείων διέλευσης και των συνόρων είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή σύμφωνα με τη δική μου κρίση είναι θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε κατά την άποψή μου. Θα πρέπει λοιπόν να προστιμαστούμε για ε, μια τέτοιου είδου ανάπτυξη τέτοιες δραστηριότητες. Παρακολουθούμε τους σύνεγγες τι σημαίνει και τελικά πρέπει να πω ότι καταβάλουμε πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε, όπως σας είπα, να ιδρύσουμε αυτό το κέντρο κατάρτισης ε, της ε, αστυνομίας της Ιεριχούλ Αυτά προς το παρόν. Σταματάω εδώ πρόεδρε και περιμένω ερωτήσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας τους τρεις για την παρουσίαση που κάνετε και για τις εξηγήσεις που δώσατε. Έχω εγώ αρκετέ ερωτήσει να υποβάλω, υποθέτω όμω ότι και οι συνάδελφοι θέλουν να σα κάνουν ερωτήσει. Η πρώτη μου ερώτηση είναι και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εσείς αναφέρατε κύριε γνωστά στα τελευταίες παρατηρήσεις. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μία μοναδική αποστολή για όλους αυτούς τους τομείς δραστηριοτήτων. Αστυνομία, τελωνιακά θέματα, διότι θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο αποστολών που αναπτύσσονται σε μία τόσο μικρή γεωγραφική περιοχή. Ε, Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε εσείς να ενεργείτε ε, από κοινού όσον αφορά την UBAM. Θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στην ε, ε, σαφή ορισμό αυτού που είπατε ότι είστε stand-by σε ετοιμότητα. Έχετε 13 άτομα στο προσωπικό σας, είστε έτοιμοι και προσπαθείτε προσπαθείτε να προετοιμάσετε την κατάσταση όταν οριμάσει η κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό για σας, δεδομένου ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη περιοχή και ευαίσθητα θέματα. Πού ακριβώς είστε και πού θα δραστηριοποιηθείτε. Επίσης, όσον αφορά την παραστηριοποίηση της UBAM, πρόσφατες εξελίξεις με το θέμα αυτό του στολίσκου που δεν μπόρεσε να φτάσει και του μπλοκαρίσματος της Γάζα. Τι σήμαινε συγκεκριμένα για την Ούμπαμ. Σας ζήτησαν να δείτε ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν για να μπορέσει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως να αναπτύξει διάφορες αποστολές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ε, τουλάχιστον εν μέρη άρση αυτού του ε, μπλοκαρίσματος όλης περιοχής. Εκτός από το σημείο διέρευσης Ράφα θα μπορούσατε στο Αρελ και στο Καρμίς άλλα σημεία διέρευσης που αναφέρετε να δραστηριοποιηθείτε. Όσον αφορά τη Γιούπολ Κόψ, ακούγοντάς σας, κύριε Δαμιστέχο, την ίδια εντύπωση με αυτή που σχημάτισα για την ε, αποστολή του Αφγανιστάν. Θα πρέπει να υπάρχει βεβαίως ε, στρατηγική βάση στα θα προχωρήσετε, αλλά όχι επιχειρησιακές ε, δραστηριότητες. Και ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και με την είπα. Μου είπαν επίσης ότι η συνεισφορά μας είναι μόνο 400 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα το οποίο είναι ε, πολύ περιορισμένης εμβέλεια σχέδιο. Πώς βλέπετε λοιπόν ε, τα πράγματα. Πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο να βοηθήσετε τις επιχειρήσεις ανάγκες των Παλαιστινίων και με ποιο τρόπο. Και αναφέρατε Επίσης δραστηριότητες ε, που αναπτύσσετε στον τομέα της ε, υποβοήθειας κράτους σε τα κράτη δικαίου. Έχετε ε, το κατάλληλο προσωπικό προβλέπετε κάτι τέτοιο, διότι εμείς όπως ξέρετε έχουμε δυσκολίες κυρίως με, την, με καλά καταρτισμένο προσωπικό σε θέματα νομικών, δικαστών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ο κύριος Κουαλτιέρη θέλει το λόγο. Grazie eh, Presidente, io ringrazio Rompenhauer Ευχαριστώ Πρόεδρε. Per la loro presenza qui e per Και για τους δύο επικεφαλείς ε, των αποστολών που εκπροσωπούνται θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον ε, και σε Κλόμπενχάουερ για την παρουσίασή του. Μας παρουσιάσατε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο αποστολές σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία οι αποστολές αυτές και θεωρώ ότι η UBOM και η UPOL δεν ε, συγκαταλέγονται στις αποστολές εκείνες όπου θα πρέπει να γίνουν περικοπές. Αντιθέτως, θα πρέπει αντιθέτως να ε, επενδυθούν πιο πολλά στις αποστολές αυτές. Και αυτό αφορά και τις προβληματικές σχέσεις ε, ως προς την ερνευτική διαδικασία, αλλά αυτό που λείπει είναι και σωστός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων μέσων που διαθέτει η ευρωπαϊκή πολιτική. Τα προβλήματα αυτά όμως θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μια συνολική μεγαλύτερη δέσμευση στην Παλαιστίνη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έπρεπε να οδηγήσει στην αναβάθμιση των δύο αυτών αποστολών. Ο κύριος Πρόεδρος έχει θίξει, ήδη πολύ σημαντικά στοιχεία να κάνω λοιπόν και μία ερώτηση παραπάνω σε ό,τι αφορά ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ό,τι αφορά, αφορά το γεωπολικό. Θα ήθελα να ρωτήσω αναφορικά με το ρόλο της πολιτικής αστυνομίας και σε ό,τι αφορά την ε, διάδοση των διαφόρων συσκευών ασφάλειας. Το γεγονός ότι θα πρέπει να μπορεί να επιβληθεί η αστυνομία δεν αποτελεί μόνο ένα από τους στόχους της αποστολής. Θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό καταβάλλονται διπλωματικές ε, προσπάθειες εκ μέρους της Ευρώπης και κατά πόσο μπορούν να βελτιώσουν αυτές οι προσπάθειες τον ρόλο της αστυνομίας. Άρα, από, πολιτικό, από πολιτική σκοπιά, τι γίνεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν γίνεται οτιδήποτε, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις με την Green Force και με τις άλλες ε, δυνάμεις στο εσωτερικό του Παλαιθνιακού Μηχανισμού Ασφαλείας και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των αποστολών. Εγώ προσωπικά είμαι απόλυτα σύμφωνος, αλλά θα ήθελα από πρακτικής άποψης να με ενημερώσετε πού βρισκόμαστε στην τρέχουσα ε, διαδικασία και πώς ε, το εκτιμούμε το θέμα και από δημοσιονομικής πλευράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πρόεδρος, η κυρία Νέιτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ τους κυρίους για τους απολογισμούς που κατέθεσαν εδώ. Κάποιοι από τους συναδέλφους ε, αναφέρθηκαν στο ότι το μεθοριακό φυλάκιο της Ράφα είχε κλείσει μετά από την ανάλυψη του ελέγχου από την Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας. Έτσι είπατε. Δεν ε, βάλω καθόλου για την ακρίβεια της δήλωσης, αλλά τα πράγματα δεν είναι λίγο πιο σύνθετα από αυτό. Δηλαδή, έκλεισε το φυλάκιο, παρέμεινε κλειστό. Αυτό δεν οφείλεται σε μια πληθώρα αιτίων πέρα από την ανάληψη του ελέγχου της περιοχής από την Χαμάς. Αυτό ισχύει, αλλά συνδράμουν και άλλες αιτίες. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο περισσότερο για το θέμα. Όσον αφορά τώρα την Παλαιστινική αστυνομία και τις σχετικές προσπάθειες, ε, η ερώτηση μου είναι η εξής. Πιστεύετε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δικαιολογεί την απαγόρευση των περιπολιών τους εκ μέρους του Ισραήλ. Η μπορεί να ξαναδιδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά στην περιοχή. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Σε κάποια φάση η Αίγυπτος, αν δεν κάνω λάθος, μονομερός άνοιξε τα σύνορα από την δική της πλευρά, δεν ξέρω αν αυτό συνεχίζει να ισχύει, υποσχόμενοι ταυτόχρονα να καταστρέψουν τις υπόγειες σύραγγες. Τι γίνεται με αυτό, γιατί όσο υπάρχουν υπόγειες σύραγγες που διευκολύνουν το λαθρεμπόριο αλλά και την παράνομη μεταφορά οπλισμού για επιθέσεις κατά του Ισραήλ, εννοείται ότι το Ισραήλ όχι μόνο θα είναι κανοποιημένο, αλλά θα είναι σίγουρο ότι πραγματική αστυνομεύση δεν γίνεται. Κύριε μάλκουε το θέμα το νομικό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στα παλαιστινιακά εδάφη. Ακούμε όμω πολλά για συνοπτικέ δικαιέ α πούμε, στην ε, ρολίδα τη Γάζα, όπου ισχύει ε, ουσιαστικά μια μορφή της σαρίας και κάτι άλλο το οποίο γνωρίζω από το παρελθόν το θέμα της διαφθοράς στα ανώτερα επίπεδα των Παλαιστινίων ισχύει το πρόβλημα και η εντολή σας συμπεριλαμβάνει την διερεύνηση αυτών των υποθέσεων διαφθοράς καθώς και την κατάχρηση κονδυλίων τα οποία μαζικά δίνονται στους Παλαιστινίους και τα και τα οποία πηγαίνουν εκεί που δεν θα πρέπει να πηγαίνουν. Κύριε Γκόμες, κύριε Πρόεδρε, θα είχα θέσει και εγώ τα ίδια ερωτήματα λίγο πολύ. Και κύριε, αυτό το που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, ποιος είναι ο στρατηγικός αντίκτυπος, ο πραγματικός αντίκτυπος αυτού του κλιμακίου στην περιοχή. Και πώς συνδυάζεται όλη αυτή η υπόθεση με την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Να ρωτήσω μας τον κύριο Φωζερά. Είπατε κάτι για τον στολίσκο και την ε, ενδεχόμενη παρέμβαση της αστυνομίας κλπ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο από την Παλαιστινιακή πλευρά. Ε, για πείτε μας λίγο περισσότερα. Τι ακριβώς εννοούσατε όταν αναφερθήκατε στον Στολίσκο και τον ε, ενδεχόμενο ρόλο που θα έχει να διαδραματίσει η μεθοριακή Παλαιστινιακή αστυνομία και τι θα έκανε η σε αυτήν την περίπτωση. Και κάτι άλλο. Όταν αυτές οι δύο δυνάμεις δημιουργήθηκαν περί τα τέλη του 2005, μία υπόθεση που ενδιαφέρει πολύ τον κύριο Σολάνα ήταν το να συμμετάσχουν γυναίκες στην δύναμη αυτή. Μάλιστα είχε σκοπό να αναθέσει την ηγεσία μίας εκ των δύο δυνάμεων σε γυναίκα. Όχι απλώς για λόγους ισότητας, αλλά για να είναι πιο αποτελεσματικές και οι δύο δυνάμεις. Οπότε πείτε μας, σας παρακαλώ, λειτουργεί αυτό στην πράξη ή όχι. Ο κ. Μάλκουιστ είπε ότι το θέμα των ε, δύο φίλων ε, μας αφορά σε κάθε τομέα δραστηριότητα, αλλά η ερώτηση μου είναι επειδή στην περιοχή γίνονται και τα λεγόμενα εγκλήματα τιμής εντός της Παλαιστινιακής κοινωνίας επίσης λόγω του ότι την ε, λωρίδα της Γάζας διφενεύει η Χαμάς, τα πράγματα θα μπορούσαν ε, να επιδροθούν ακόμη περισσότερο. Οπότε, λείπετε μας λίγο για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Η πρώτη ερώτηση υπησέρχεται το δικαστικό ευρωπαϊκό σύστημα στις Παλαιστινιακές, ε, στα Παλαιστινιακά εδάφη ή υποβοηθάται ουσιαστικά το ήδη υφιστάμενο σύστημα το οποίο υποθέτω ότι είναι αγγλικό από ιστορικής άποψης και κατά δεύτερον ποιες είναι οι σχέσεις σας με τη Χαμάς επιτόπου. Ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαπραγματεύεται με τη Χαμάς, αλλά προφανώς πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση, κάποια επαφή για επιχειρησιακούς σκοπούς και αυτό αποτελεί πρόκληση μεγάλη. Ευχαριστώ. Κύριε Σκλομπανάουρ, έχει το λόγο. Thank you. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με τις πιο γενικές ερωτήσεις. ο ύπατος ε, εκπρόσωπος ε, εξετάζει τα θέματα αυτά πάρα πολύ ε, ενδελεχώς για να καταλήξουμε σε μια πιο ενεργή προσέγγιση. Αυτή έχει η κατάσταση επί του παρόντος. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες, καθότι δεν έχουν ακόμα δημορφωθεί. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε ε, κατάσταση, σε ό,τι αφορά τη Γάζα συγκεκριμένα. Φυσικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ πολύ σύνθετη. Το γεγονός ότι η Χαμάς είναι στη Γάζα περιπλέκει τα πράγματα, αλλά σωστά είπατε δεν είναι το μόνο που περιπλέκει την κατάσταση. Υπάρχει και άλλα θέματα, η αδυναμία των ε, Παλαιστινιακών αρχών να παρευρίσκονται στην Γάζα, στην παρούσα φάση. Και αυτό έχει να κάνει με την δικασία επανασυμφιλίωσης, η οποία ακόμα δεν έχει καταλήξει σε αυτά αποτελέσματα. Άρα, είναι πολύ σύνθετη πραγματικά η κατάσταση. Δεν είναι απλό να πούμε ότι θα περάσουμε στο ψητό κατευθείαν, γιατί υπάρχουν ακριβώς όλοι αυτοί οι παράγοντες που περιπλέκουν την κατάσταση. Εξετάζουμε λοιπόν μια βαθμιαία προσέγγιση, η οποία φυσικά προϋποθέτει πολιτική συμφωνία από πλευρά της κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής ασφαλώ Αυτό κατά πρώτον σε ό,τι αφορά την Upol Cops τώρα. Νομίζω ότι η κατάσταση στο σημείο αυτό είναι πιο ξεκάθαρη. Όλα τα μέρη συμφωνούν, θεωρώ, για το θετικό αντίκτυπο της επιχείρησης, ότι συμβάλλει στην ασφάλεια στην Βυτική Όχθη του Ισραήλ, αλλά και των Παλαιστινίων πολιτών. Με μια αστυνομία η οποία ανταπεξέρχεται καλύτερα στις προκλήσεις τις σημερινές αληθεύει ότι είμαστε παρόντες σε στρατηγικό επίπεδο. Αυξήσαμε την παρουσία μας, όπως είπε και ο συνάδελφος. Έχουμε πλέον ε, στενές εταιρικέ σχέσεις και με την Υπουργό Εσωτερικών Δικαιοσύνης, ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι αυτοί φυσικά συμμετέχουν στην κατάρτιση των προγραμμάτων ασφαλείας και σε δεύτερη φάση ενδεχομένως να περάσουμε και σε πιο επιχειρησιακό επίπεδο για να απαντήσω σε αυτό που ρώτησε ο Πρόεδρος, αλλά αυτό σε επόμενη φάση, όχι ακόμη. Θα πρέπει σε παρούσα φάση να ενισχύσουμε την παρουσία μας σε στρατηγικό ε, επίπεδο και νομίζω ότι οι επικεφαλής των αποστολών αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα σχέδια που έχουν καταστρωθεί ως προς αυτό. Ο αρμοστής ε, Μάλκβες θα αναφερθεί στο είδος της αστυνόμευσης που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Δεν θέλουμε να εξάγουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο, αν και κοιτώντας το απ' έξω, ουσιαστικά τα συστήματα αστυνόμευσης, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον παρόμοια. Δεν ε, είναι τα ίδια, αλλά είναι παρόμοια. Δεν διαφέρουν τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει, όσο τα συστήματα αστυνόμευσης ε, της Μέσης Ανατολής. Μας απασχολεί πολύ το θέμα της αποτελεσματικότητας και ως τώρα έχουμε δει ότι υπάρχει θετικός αντίκτυπος από τις δύο αποστολές. Είναι πολύ συγκεκριμένη η αποστολή τους. Δεν θέλουμε να περιπλέξουμε τα πράγματα. Αναμειγνύοντας, αν θέλετε, για παράδειγμα, τους πόρους των δύο αποστολών. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό εξαρτάται φυσικά από το ευρύτερο πλαίσιο και από το στόχο που επιδιώκουμε. Η επικεφαλής ε, των αποστολών, επικεφαλής ε, της αποστολής COPS θα σας μιλήσει πιο μωρό... σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της αποστολής του, αλλά δεν νομίζω ότι τύφεται θέμα λογοδοσίας, ε, ο στρατηγικός αντικτύπος τώρα. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Είναι σημαντικό μάλλον να αντιληφθούμε ότι η εντολή μας περιορίζεται στην μη στρατιωτική αστυνόμευση και μιλάμε για το, την πράσινη αστυνόμευση. Εμείς, οι Αμερικανοί μάλλον, ε, εστιάζονται στο green policing. Εμείς ε, εστιαζόμαστε στην πολιτική αστυνόμευση. Ίσως να μην είναι τόσο εντυπωσιακό το σκέλος αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και σημαντικό για τους Παλαιστινίους, γιατί βελτιώνεται η ασφάλεια στον δρόμο και επίσης περιορίζονται και τα περιθώρια ακραίων ε, φαινομένων. Πρόκειται για μια προσέγγιση λιγότερο εντυπωσιακή ίσως, αλλά εξίσου σημαντική θεωρούμε για το θέμα τώρα της ευκρίνεια της αποστολή Από δική μας ε, πολιτικής άποψης υπάρχει επιθυμία να υπάρχει τέτοια προβολή. Αλλά παράλληλα μας αποσχολούν πάρα πολύ τα θέματα και οι αρχές της ιδιοκτησίας. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα έχει και τα δύο για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Είναι σημαντικό να μην, είμαστε, να μην προβαλόμαστε ιδιαίτερα, να θεωρούνται ότι είναι δικές του οι δυνάμεις και να μην φαινόμαστε ότι εμείς ερχόμαστε να επιβάλλουμε το οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν κρατούμε χαμηλό προφίλ όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και όντω, αυτό περιορίζει κάπω ε, την προβολή των δυνάμεών μα. Αλλά αυτό είναι το τίμημα το οποίο θα πρέπει να πληρώσουμε, γιατί προτιμούμε να κρατήσουμε την αρχή τη ιδιοκτησία, αν θέλετε, την αρχή τη ε, ανεξαρτησία. Επειδή λοιπόν τηρούμε χαμηλό προφίλ και επειδή ε, η αποστολή μας είναι λιγότερο εντυπωσιακή, Μπορεί να έχετε την εντύπωση ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική, αλλά θεωρούμε ότι συμβάλλει πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά το μέλλον τώρα, θεωρώ είναι πολύ ασταθές το πολιτικό συγκείμενο στο οποίο λειτουργούμε. Δεν θέλω λοιπόν να προκαταβάλω το οτιδήποτε. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια καλή βάση επί της οποίας μπορούμε να συνεχίσουμε. Και τα υπόλοιπα ερωτήματα να τα απαντήσουν οι επικεφαλής των αποστολών. ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το ε, θέμα της μη αποστολής, δεν απαντήσω, απέντησε ο ΚΕΣ. Όσον αφορά την δραστηριότητα σε καθημερινή βάση που αναπτύσσουμε, πρέπει να σας πω ότι πάντα προετοιμάζουμε την μελλοντική μας ανάπτυξη και είμαστε και σε επίπεδο εξοπλισμού, οχημάτων και σε προσωπικό επίπεδο πάντα έτοιμοι και ίσως ξέρετε ότι στο παρελθόν μέναμε σε ένα ξενοδοχείο. Τώρα είμαστε σε ένα αρχηγείο, αν θέλετε, πιο αποδεκτό. Και Επίσης πρέπει να πω ότι μπορέσαμε και με τα κονδύλια που είχαμε να αγοράσουμε τα οχήματα που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να ενεργούμε αποτελεσματικά. Διότι στο παρελθόν η Ιταλία μας παρήχε το μεγαλύτερο ποσοστό των μέσων που είχαμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, χάρη στην δουλειά αυτή που κάνουμε σε καθημερινή κάθε, είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε το σύνολο των δυνάμεων που διαθέτουμε σε τρει εβδομάδε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε αμέσως. Βεβαίως δεν ε, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτή την ε, διοικητική και υποστηρίξη ε, δραστηριότητα μόνο. Θέλουμε να επιδείξουμε και το ενδιαφέρον που έχουμε για όλη τη διαδικασία ειρήνευσης και για να μπορέσουν να επωφεληθούν όλοι από τις γνώσεις μας και την προγραμματογνωσία πρέπει να σας πω ότι το θέμα της πραγματογνωμοσύνης των ε, γνώσεων που διαθέτουμε είναι κάτι το οποίο τη χάνει γενικότερης αποδοχής από όλους. Τι είπα, όλες τις διεθνείς οργανώσεις, όλους τους εταίρους που αναγνωρίζουν και έρχονται συχνά στη Γιούμπαν για να μπορέσουν να συναντήσουν τους υπεύθυνους διαχείρισης συνόρων τελων... θέματων που αφορούν τα τελωνία και παρέχουμε σε όλους του ενδιαφερόμενου. με Αμερικανούς ε, εταίρους, με ε, συναδέλφους της Πολκόψ, συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας για να επωφεληθούν οι Παλαιστίνοι από αυτή την πραγματογνωμοσύνη, λέω. Η πιο σημαντική μας δραστηριότητα είναι ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός. Δηλαδή, κάθε φορά που βλέπουμε να υπάρχει κάποια ακτίδα κάποια ελπίδα όταν λέγεται ότι υπάρχει περίπτωση Παλαιστίνη να μπορέσουν να αναπτύξουν μια πολιτική ανοίγματο συμφιλίωσης. Παρεμβαίνουμε. Ίσως προηγουμένως δεν εκφράστηκε σωστά για τον Στολίσκο. Αυτό θέλω να πω. Μόλις ακούσαμε ότι είπε είπε ότι οι εκπρόσωποι θα πρέπει να ανοίξουν τα σημεία διέλευσης, να διευκολυνθεί η κατάσταση αμέσως αρχίσαμε να δουλεύουμε και με τις γνώσεις που έχουμε επί διότι ξέρουμε πώς λειτουργούν όλα τα σημεία διέλευσης, υποβάλαμε προτάσεις στο στρατηγείο για να επιληθεί το πρόβλημα. Καθημερινά, λοιπόν, προσπαθούμε να ε, κάνουμε κάτι χρήσιμο μην πιστεύετε ότι καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Ίσως ορισμένοι έχουν εδώ αυτήν την άποψη, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Αυτό, αυτή είναι η απάντηση που θέλω να δώσω για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο σταματήσαμε τις δραστηριότητες μας στη Ράφα, ο κύριος λόγος, ο επίσημος, είναι ότι όντως η παρουσία της Χαμάς κατά κάποιο τρόπο απο, ε, μας υποχρέωσε διότι από τα θέματα τακτικής και πολιτικής δεν μπορούσαμε να σε συνομιλία μαζί τους και πρέπει να πω ότι αυτό το γεγονός προκάλεσε και κάποιες άλλες αντιδράσεις, αμέσως αντέδρασε το Ισραήλ, το οποίο πολλές φορές για λόγους ασφαλείας βάζει κάποια τροχοπέδη στις δραστηριότητές μας. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, αρχίζουν να επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους ενέργειες. Και είπε ο συνάδελφος ότι κάποιες φιξέλες πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσουν οι δραστηριότητές μας. Αν θέλετε λοιπόν να σας πω ότι όλα αυτά έγιναν μετά από την ανάληψη της Χαμάς, το λέω. Όσον αφορά το ρόλο της Αιγύπτου άνοιγμα ή όχι του σημείου διέλευσης Ράφα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες η ασφάλεια για να καταστήσει ασφαλή αυτή την περιοχή, υπάρξει ένα ε, υπόγειο στίχος για να μπλοκάρονται τα τούνελ μεταξύ των αστυνομικών και των τελωνοφυλάκων στα σύνορα υπάρχουν δράσεις των Αιγυπτίων για να μειωθεί ο ρυθμός των ε, τούνελ, οι Ισραηλινοί επίσης τελείωσαν την δουλειά βομβαρδίζοντας, άρα μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των τούνελ. Μιλούσαμε για χιλιάδες και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για 400, τα οποία σιγά σιγά μειώνονται σε 100. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται πιο ασφαλής η περιοχή. Και βεβαίως αποτελούν τα τούνελ σημείο ανασφάλειας για τους Ισραηλινούς. Σας είπα επίσης τι έγινε με τον Στολίσκο. Προσπαθήσαμε όλες τις πληροφορίες που είχαμε επιτόπου να τις διαβιβάσουμε και βεβαίως ασχολούμεθα και με το θέμα των δυνατοτήτων να ξανανοίξει. Τώρα, όσον αφορά το περίφημο gender, την ε, ε, ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Προσπαθούμε πάντα να το σεβόμεθα. Αυτό ως αρχή. Βεβαίως, θέλουμε και εμείς να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δεν είχε γυναίκες στα σημεία διέλευση. Ζητήσαμε επίσης να υπάρχουν γυναίκες. Επίσης στην ε, επιχείρηση κασλέντ. αναπτύξαμε 45 άτομα, 10 από τα οποία είναι γυναίκες. Και τώρα έχουμε 13 άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων 3 είναι γυναίκες. Αυτό το λέγω για το gender equilibrium. Ευχαριστώ. Ελπίζω να πάτε στις ερωτήσεις σας. Ε, um, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επαντήσω ως προς τον στρατηγικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας. Συγγνώμη, δεν ήμουν αρκετά σαφής. Φαίνεται, έδωσε την εντύπωση ότι δεν έχουμε επιχειρησιακό ρόλο στην περιοχή. Και όμως, Προσέξτε, επειδή κάποιοι είπαν κάτι σχετικό, άλλο Αφγανιστάν, άλλο Παλαιστίνη. Έχουμε αστυνομία, έχουμε εισαγγελεί, έχουμε δικαστές, έχουμε ένα σύστημα. Έχει πολύ μεγάλε ελλείψει, αλλά υπάρχει το σύστημα και λειτουργεί. Στο παρελθόν, 2005, 2006, 2007, το κλιμάκιο είχε επιχειρησιακές δραστηριότητες στην τελική όχθη στην Λωρίδα της Γάζας, όχι πια τώρα βεβαίως. Είχαμε πάντοτε πρόσβαση στα στελέχη της αστυνομία στην περιοχή. Κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Συνεχίσουμε τις επισκέψεις κάθε εβδομάδα. Όταν ανέλαβα πάντως τα καθηκοντά μου φέτος, πριν από μερικούς μήνες, ε, σχημάτισα αμέσως την εντύπωση ότι μάλλον γίνονταν υπερβολικά πολλές Γι' αυτό καθέρωσε ένα πρόγραμμα βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση του προσωπικού έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετοί και επιτόπου έξω και οι επιχειρήσεις όπως λέμε και στα γραφεία για να υποστηρίξουμε ακριβώς τα στρατηγικά σχέδια που έχουμε καταστρώσει. Έτσι θα επιτευχθεί η συνεργεία. Φαίνεται ότι αυτή η λύση είναι καλή και αποδοτική. Αναδιοργανώσαμε λοιπόν λίγο. Είμαστε στην περιοχή κάθε εβδομάδα και θα επανέλθουμε με ενισχυμένες δραστηριότητες. Αυτό είναι τουλάχιστον το πρόγραμμα, ο σκοπός μας. Και κάτι άλλο, όλα αυτά αναγνωρίζονται και από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Αν έχουμε επαρκε προσωπικό τώρα. Ναι, για το συγκεκριμένο κλιμάκιο. Ναι, είμαστε σε καλή θέση και αρκούμε και όταν, για τις περιπτώσεις που μας καλούν τις αποστολές της ε, Μπορεί να μην ισχύει αυτό για όλες ε, τις περιπτώσεις, αλλά γενικά είμαστε αρκετοί. Τι είδους επίσης δραστηριότητες μπορούμε να υποβοηθήσουμε. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον άλλο ερώτημα. Εγώ συναντώ τακτικός, όπως είπα, με τους ε, Παλαιστινίους για να έχουμε και καλές διπλωματικές επαφές και φυσικά αναφέρομαι σε διαβάσεις τους του μου στις Βρυξέλλες. Σίγουρα μπορούν να γίνουν περισσότερα και μπορώ να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή οι Παλαιστίνοι είναι έτοιμοι να λάβουν την ευθύνη για την ανάπτυξη και την ασφάλεια μιας ολόκληρης περιοχής. Στην περίπτωση αυτή που προχωρήσουν τα πράγματα θα μπορούσαμε να περάσουμε εκπαίδευση για υποδομές έτσι ώστε να διασφαλιστούν και να προστατευτούν αυτές οι περιοχές. Η οικονομική κατάσταση δεν είναι κακή, είναι ικανοποιητική. Για να καλύψουμε τα έξοδα του 2010 χρειαζόμαστε μία μικρή μόνο ένεση, την οποία ήδη έχουν εγκρινεί οι επιτροπέ. Για το 2011 καταρτίζουμε τώρα τον προπολογισμό και φαίνεται ότι ο προπολογισμό θα καλύψει σχετικά άνετα τι δραστηριότητέ μα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά άτυπα τουλάχιστον μπορώ να σα πω ότι τα πράγματα είναι σε καλή κατάσταση. Όσον αφορά τι ε, βραδινέ νυχτερινέ περιπολίε, είναι όντω Όντως σε ορισμένε περιοχέ, δεν έχει την άδεια η Παλαιστινική αστυνομία να περιπολεί, το οποίο είναι κρίμα. Και όχι μόνο για την PCP. Το γενικότερο πρόβλημα είναι ότι αφαιρείται έτσι νομιμοποίηση από την αστυνομία αυτή, όταν μάλιστα εισβάλλουν οι σελήνοι. Και το είπα αυτός τους Ισραηλινούς συνομιλητές μου. Μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση αυτή η ιστορία. Και όπως είπα στην εισαγωγή μου, αν θέλουμε να σημειώνουμε πρώτα στην περιοχή, χρειαζόμαστε νομιμοποίηση. Τώρα για, την ε, συνοπτική, για τις συνοπτικές δίκες στη Γάζα δεν μπορώ να απαντήσω, δεν πηγαίνω, δεν ξέρω. Απλώς δεν ξέρω και δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Όσον αφορά την διαφθορά τώρα, δεν έχουμε σχετική εντολή διερεύνησης των φαινομένων διαφθορά. Παρέχουμε συμβουλευτική καθοδήγηση και ω εκεί. Εκπαιδεύουμε όμως εισαγγελεί και δικαστές για το θέμα. Πρόσφατα μάλιστα βοηθήσαμε την ίδρυση ενός σχετικού σώματος, το οποίο είχαμε συζητήσει πρόσφατα. Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό στο ανώτερο δηλαδή επίπεδο. Είναι μια πρωτοβουλία που υποστηρίζουμε σε μεγάλη έκταση και μάλιστα έντονα. Αυτή τη στιγμή 67% του στελεχικού μας δυναμικού είναι γυναίκες. Δεν μπορούσε να είναι περισσότερο κυρίως στα ανώτερα κλιμάκια. Διότι στα ανώτερα κλιμάκια υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες. Θα προσπαθήσουν να έρθουν και άλλες γυναίκες να λάβουν ανώτατες θέσεις, δύσκολο όμως, γιατί υπάρχουν λίγες εκπαιδευμένε γυναίκες που κάνουν αίτηση. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε σε συνεργασία και με τα κρατημέλη. Να αναδειχθούν δηλαδή καλές γυναίκες υποψήφοι. Ως προς τη Σουηδία, ξέρω ότι υπάρχουν πολύ καλές ε, Σουηδέζες και πιστεύω ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει, να συμμετάσχουν τελικώ περισσότερες γυναίκες στην Παλαιστινιακή αστυνομία. για το θέμα τη ισότητα των δύο φύλων, εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβαίω, ναι. Η άλλη ερώτηση αφορούσε Εάν ε, εμπλεκόμαστε σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων μας. Καταρχήν αυτό συμβαίνει στην εκπαίδευση και το προσπαθούμε. Επίσης με την ε, Παλαιστινική αστυνομία καταρτήσαμε ένα μοντέλο, ας το πω έτσι, για να συζητήσουμε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου. και επίση δημιουργήθηκε ένα γραφείο παραπώνων σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Επιτροπή με τον Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Εγώ είμαι επικεφαλής της ε, αποστολής πάντως παρακολουθώ οτιδήποτε ακουστή που μπορεί να έχει σχέση με την αποστολή μα που συμπεριλαμβάνει και τα δικαιώματα του ανθρώπου και αν η υπόθεση έχει κάποιες απαιτήσει θα συμβουλευτώ. Παντώ Πάντως, σε κάθε περίπτωση θεσπίζουμε μηχανισμούς επιτήρησης ελέγχου της Παλαιστινικής αστυνομίας, στην προσπάθειά μας να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθούμε. Το τι αστυνομικό μοντέλο εφαρμόζουμε. Όπως είπε ο κ. Κοπενχάουερ, δεν υπάρχει ένα, αλλά περισσότερα μοντέλα. Άλλωστε στοιχεία έχουμε πάρει και από τους Ισραηλινούς. Σε μερικές περιπτώσεις, σε υποθέσεις με τεχνικές απαιτήσει. Δηλώνωσαμε εκπαιδεύσεις Και έχουμε μάλιστα και στο Τελαβίβ ε, ε, ένα αστυνομικό υποτμήμα. Εφαρμόζουμε επίση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα με βάση φυσικά τι δυνατότητε στην περιοχή, με τα μέσα που έχουν οι Παλαιστίνοι. Σε ορισμένε περιπτώσει χρειάζεται να ζητήσουμε κάτι από τα γειτονικά αραβικά κράτη. Καμιά φορά όμω στρέφουμε και αλλού, α πούμε, στι ευρωπαϊκέ χώρε, το μοντέλο αυτό είναι λίγο πολύ το ίδιο, όπως ας πούμε στην ε, σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, στην, όπω είπα, προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τώρα για τη Χαμάς, Δεν έχω να πω πολλά για την Χαμάς, γιατί δεν έχω επαφέ με την Χαμάς στην περιοχή, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω. Να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να παραλύσω το Αφγανιστάν με την Παλαιστίνη. Εννοείται ότι ε, δεν είναι συγκρίσιμε οι δύο περιοχέ. Απλώ στα πλαίσια τη ΚΕΠΑ πάντα διερωτώμεθα ποιο είναι ο στρατηγικό αντίκτυπος. Διερωτώμεθα αν ο συνδυασμό μα αποδίδει γι' αυτό και αναφέρθηκα στο τακτικό ή επιχειρησιακό επίπεδο Κατανοώ ε, φυσικά τη διαφορά μεταξύ αυτών που κάνουμε με τους Αμερικανούς, με την γαλάζια, την πράσινη αστυνομία. Αλλά εμείς, σε κάθε περίπτωση, οι Ευρωπαίοι, για τους σκοπούς της διατήρησης της ε, τάξης, για τις ε, μεν τις επιχειρήσεις με τους Γάλλους τους Ιταλούς. Λείπουμε κάπως, αν θέλετε, από, τη, από το σκηνικό, ενώ έχουμε τεχνογνωσία. Η κυρία Νικολάη, πρόεδρε, δύο ερωτήσει. Πολύ συγκεκριμένα. Ο ποινικό κώδικα στην περιοχή προβλέπει ακόμη την ποινή του θανάτου. Η Χαμάς ε, ενέκρινε ποινές, θανατικές ποινές. Και το δεύτερο ερώτημα έχει σχέση με την συμπεριφορά του Ισραήλ. Ποιες είναι οι συνθήκες διοικητικής κράτησης. Πρόκειται για την εντολή, την απόφαση του 2007 που επιτρέπει την προσωρινή κράτηση, επί ένα εξάμεινο μάλιστα. Ε, ισχύουν αυτά ακόμη στην περιοχή. Κύριος Φάγκελ. Η δική μου ερώτηση είναι ακριβώς η ίδια ή περίπου μάλλον η ίδια. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποιες οι σχέσεις σας ε, και έχετε μάλλον σχέσεις εργασίας με τους θεσμούς των Ισραηλινών, με τις αρχές, τις Ισραηλινές, με την αστυνομία. Πώς τοποθετούνται απέναντι σε αυτά που κάνετε. Εκτιμούν τις προσπάθειές σας. Θέλουν να γυρίσετε να πάτε σπίτια σας. Και πώς αισθάνεστε εσείς, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την αποστολή σας ως προς τον πολιτικό στόχο που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη, δηλαδή την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών. Προφανώς εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου όλο και πιο λίγα γίνονται και όλο πιο περιορισμένη είναι η βάση για μια λύση δύο κρατών. Φαίνεται ότι όλο και πιο πολύ περιορίζεται το περιθώριο για τη λύση αυτή των δύο κρατών. Όταν λοιπόν θα ολοκληρώσετε την εκπαίδευση των Ισραηλινών αστυνομικών, τι θα κάνουν οι αστυνομικοί αυτοί. Είναι μάλλον ε, απεσιόδοξη η πλευρά μου που παρουσιάζω και η ερώτηση που θέτω και θα ήθελα να ακούσω μια ειλικρινή απάντηση εκ μέρου σα. Ευχαριστώ, κύριε Χάουρθ... Να απαντήσει για τον ποινικό κώδικο, κώδικα ο αρμοστή ε, Μάλλον Κουβέστη, γιατί δεν είναι δικό μου τομέα, για την πιο πολιτική ερώτηση για τη λύση των δύο κρατών. Αναφέρθηκα σε αυτό γιατί πρόκειται για μια δεδηλωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης τόνισα ότι Θεωρώ ότι η αποστολή η COPS ε, συμβάλλει στην ασφάλεια επιτόπου και αυτό από μόνα του ευνοεί την ασφάλεια και την σταθερότητα. Και την όλη πολιτική διαδικασία ασφαλώς, χωρίς να προδικάζω ασφαλώς το αποτέλεσμα της ε, πολιτικής αυτής διαδικασίας. Το τόνισα αυτό από τις επαφές μου με τις Ισραηλινές ε, αρχές και με τον Υπουργό Άμυνας μου δείχνουν ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη της ε, αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανέφερε και ο αρμοστής Μάλλον Κουβέστ σε ό,τι αφορά με τις, ε, τις επαφές του με την ε, αστυνομία επιτόπου. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι είναι θετική η στάση έναντι των όσων κάνει η Γιουπολ COPS Ασφαλώς και υπάρχουν περιορισμοί ωστόσο και τις ανέφερε και ο αρμοστής. Μίλησε για παράδειγμα για τις νυχτερινές ώρες και φυσικά υπάρχουν και γεωγραφικοί περιορισμοί. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, η ζώνη Α νομίζω αναφέρεται, όπου δρούν οι Παλαιστινιακές αρχές και κάποιες άλλες ζώνες στις οποίες δεν μπορούν να δράσουν. όσο έχουν λοιπόν τα πράγματα σήμερα, η αρρωγή μας περιορίζεται στο πλαίσιο αυτό. Έχει αυτούς τους περιορισμούς, αλλά και στις ζώνες αυτές ακόμη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης από επιχειρησιακής άποψης. Και εδώ έρχεται το ερώτημα του Προέδρου. Η ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ασφαλώς και αυτή είναι η πρόθεσή μας. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει ότι θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, και η Ισραηλινή κυβέρνηση και η Παλαιστινιακή πλευρά, γιατί είναι ασφαλώς ε, ευαίσθητο το θέμα αυτό. Αλλά ως προς αυτή την άποψη θα θέλαμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αλλά θα πρέπει φυσικά σε στρατηγικό επίπεδο να υπάρχει συμφωνία για το ποια είναι τα σχέδιά μας, προς τα που οδεύουμε, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και ούτω καθεξής. Άρα, για να απαντήσω, εν συντομία, μπορεί οι συνομιλίες να είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μπορεί να είναι ευαίσθητο το πολιτικό κλίμα, Πρόκειται για ένα περιορισμό της αποστολής, αλλά ακόμα και στην κατάσταση αυτή μπορεί να συνεχίσει την εργασία της η αποστολή προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή μου. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον αρμοστή για να απαντήσει και το θέμα του ποινικού κώδικα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ποινικού κώδικα έχουμε δώσει τεχνικές ε, πληροφορίες και τεχνική αρρωγή και φυσικά ήταν μακρά η διαδικασία αυτή. Ένα πρόβλημα είναι ασφαλώς ότι δεν υπάρχει κοινοβούλιο. Και ανέφερα και χθε ότι έγινε μια συνδιάσκεψη υψηλού επίπεδου σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα με την παρουσία του κ. Φαγιάτ και η έκθεσή μου είναι ότι αναφέρθηκε στο θέμα της αντικής καταδίκης στην παρέμβαση του χτες και λίγο πολύ ανέφερε ότι με προεδρικά διάταγμα ουσιαστικά θα καταργηθεί η θαντική καταδίκη. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές πτύχες που ρωτήσατε για το Ισραήλ. Δεν γνωρίζω για τις εργασιακές μας σχέσεις τώρα με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά την αστυνομία. Συναντιέμαι τακτικά και το προσωπικό μου συναντιέται τακτικά με εκπροσώπους της Ισραηλινής ε, αστυνομίας και με το Γενικό Αρμόδιο για την ε, Δυτική Όχθη. Έχουμε τακτικές συναντήσεις, συναντιέμαι και με εκπροσώπους ε, του Υπουργείου Άμυνας και Εξωτερικών. Αυτοί είναι οι βασικοί συνομιλητές από πλευράς του Ισραήλ. Τι αναφέρουν λοιπόν, αν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε. Είναι σαφής η εντύπωσή μου ότι ναι, τους αρέσουν τα όσα κάνουμε και ότι αντιλαμβάνονται ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια και ως προς αυτό νομίζω ότι η αποστολή έχει πραγματικά συμβάλει στην βελτίωση της κατάστασης και αυτό το παραδέχονται και από Ισραηλινής πλευράς. Και μας λένε ότι θέλουν να συνεχίσουμε το έργο μας και ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Για τη λύση των δύο κρατών. Φυσικά είναι πολιτικό το θέμα αυτό, συμφωνώ. Το τι κάνουμε εμείς όμως, όπως είπε και ο κ. Κλόπενχάουρ, είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να οικοδομηθούν ισχυροί θεσμοί προκειμένου στο τέλος να καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση δύο κρατών. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, πότε είναι μάλλον η αστυνομική δύναμη, η εισαγγελία έτοιμη για να σχηματιστεί κράτος, θα απαντάει αυτό. Είναι πολιτικό θέμα, είναι πολιτική αυτή η εκτίμηση σε τελική ανάλυση, ξέρετε. Bien, s'il n'y a pas d'autres... δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι για να ολοκληρώσουν τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε τα όλα αυτά τα θέματα των ε, αποστολών στην Παλαιστίνη μετά τις παρούσες αναθεωρήσεις. Κανείς δεν θέτει ένα αμφιβόλο την ε, ανάγκη να έχουμε αποστολές επιτόπου και βεβαίως τίθεται θέμα της εντολής τους, της εμβέλειάς τους. Όπως είπατε, είναι δύσκολο από πολιτικής πλευράς το όλο εγχείρημα. Ελπίζουμε όμως ότι η εκπρόσωπος θα μας εξηγήσει πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια δύναμη πιο συνεκτική και αποτελεσματική. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Euh, και έχουμε μετά την ε, διάσκεψη του διευρυμένου προϊόντου, με τους συντονιστές. Υπενθυμίζω σε όλους ότι αύριο έχουμε το πρωί ακρόαση για την ε, αντιπυραυλική ασπίδα. Αύριο στις 9 λοιπόν.